Λοιπόν, θα προχωρήσουμε στις επεξηγήσεις ψήφου. Ο πρώτος είναι ο κύριος Μαμίκινς. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα συμφωνήσω ότι η δημοσιονομική σταθερότητα θα πρέπει να τύχει εγγυήσεων και θα πρέπει να έχει προτεραιότητα σε σχέση με άλλου είδους ε, οικονομικές καταχρηστικές λογικές. Δεν μιλάμε για ένα παιχνίδι ηλεκτρονικών υπολογιστών, γιατί σε αυτή την περίπτωση οι συνέπειες αποτυχίας ενός ε, τέτοιου επικίνδυνου παιχνιδιού είναι σημαντικές για όλους. Thank you, Ευχαριστώ συνάδελφε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την κυρία Κρούπα για ένα λεπτό. Ε, Εγώ ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος για την καταπολέμηση της παρενόχλησης όχι μόνο στον τόπο εργασίας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου υπάρχουν αντιπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Εθνών που κανονικά έχουν κάποιο, κάποιο γόητρο σε σχέση με την δραστηριότητά τους. Έχουμε συμφωνήσει λοιπόν με αρκετές ρήτρες της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και θα πρέπει να μην μειωθούν οι δράσεις μας γύρω από τον τομέα αυτό στο μέλλον. Θα πρέπει ε, να μην νομοθετούμε με τρόπο ο οποίος λειτουργεί εναντίον της έννοιας της οικογένειας, της ελευθερίας και των χριστιανικών αξιών. Δεν θα πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι το ανθρώπινο όν είναι πλήρως απελευθερωμένο από τα ίδια του τα βιολογικά χαρακτηριστικά και δεν θα πρέπει να διαφημίζουμε εναλλακτικέ μορφές ε, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού. Στο ίδιο θέμα η κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ, όπως προλαλή σας συνάδελφος, να πω ότι είναι τελείως απαράδεκτη η σεξουαλική παρενόχληση. Και συμφωνώ, όπως και άλλοι βουλευτές, ότι και ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να καταπολεμήσουμε και να εκριζώσουμε αυτή την ε, παρενόχληση. Έχω ε, επίσης προτείνει συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δυστυχώς ορισμένοι συνάδελφοι προσπάθησαν να το εκμεταλλευτούν αυτό, έτσι ώστε κάποια κράτη-μέλη να κυρώσουν τη Σύμβαση Κωνσταντινούπολης. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι υποχρέωση αυτό. Το Κοινοβούλιο δεν έχει μία αρμοδιότητα ε, να επιβάλλει οτιδήποτε στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για το ίδιο ψήφισμα. Γιουρέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και η κυρία Ζαμπόσκα θεωρώ ότι είναι σκάνδαλο να χρησιμοποιήσουμε το δράμα αυτό των γυναικών που υφίστανται επιθέσεις για να προωθήσουμε ε, κάποια πρότυπα της συμβάσεως της Κωνσταντινούπολης. Ξέρουμε τι συμβαίνει στην κινηματογραφική βιομηχανία σε σχέση ε, με την σεξουαλική αυτή ε, επίθεση την οποία υφίστανται οι γυναίκες. Δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές αυτές και στο κοινοβούλιο μας θα ήθελα λοιπόν να απαιτήσω αυτοί που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες με τέτοιο είδους απαράδεκτο τρόπο αυτοί να τους ονοματίσουμε, να τους ντροπιάσουμε. Ξέρουμε επίσης ότι οι αστυνομικές αρχές αποκρύβουν τα στοιχεία που συσχετίζουν την παράνομη μετανάστευση με τις επιθέσεις εις βάρος των γυναικών. Θα περάσουμε τώρα στις επεξηγήσεις ψήφου της εκθέσεως ΕΚΜΑΡΚ. Ο κύριος Μαμίκιν σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θέλω να υπογραμμίσω την σημασία που έχει η πολιτική συνοχής. Είναι το ισχυρότερο μέσο για την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Στην Λετωνία καλύπτει το 70% των επενδύσεων στην πολιτική της υπαίθρου. Νομίζω ότι ε, τα χρήματα μετά το 2020 δεν θα πρέπει να μειωθούν. Η Λετωνία δυστυχώς έχει χάσει το 1 τρίτο του πληθυσμού της τα τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης προοπτικών και των χαμηλών μισθών. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να μειωθούν οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγώ φυσικά υπερψήφισα την πρόταση. Ευχαριστώ συνάδελφε. Ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τσαμπάτσκι. Χωρίς μικρόφωνο ο κύριος Τσαμπάτσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ καταψήφισα την έκθεση αυτή. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία στην έκθεση τα οποία δεν μπορώ να δεχτώ. Η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι ίδια σε όλη την Ευρώπη και δεν μπορεί τα μέτρα να είναι ενιαία. Διαφωνώ λοιπόν με τις προτάσεις οι οποίες γίνονται για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας των μεταναστών. Πρώτα θα πρέπει να λύσουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα και τις τεράστιες διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πάρει κυρώσει ει βάρο των κρατών μελών που ακολουθούν προστατευτικέ πολιτικέ, όπω το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γαλλία, γιατί στην Ανατολική Ευρώπη το μέλλον της Ευρώπης οι νέοι έχουν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα στην έκθεση Κάσπαρη, διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία. Για ένα λεπτό, Σελίμοβιτς πρώτα απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Αυστραλία και η Σουηδία έχουν μεγάλη εμπορική παράδοση. Συνεργάζονται, έχουν την ίδια επιχειρηματική νοοτροπία. Κάπου χίλιες σουηδικές επιχειρήσεις ε, δραστηριοποιούνται στην Αυστραλία. Πρόκειται για 11 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες εξαγωγές της Σουηδίας προς την Αυστραλία. Οπότε Θέλω να κάνω έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους Αυστραλούς ε, εταίρους να φροντίσουν να υπάρχει διαφάνεια και να μην χρειαστεί να περιμένουμε πολύ περισσότερο μέχρι να αρχίσει να ισχύει η συμφωνία. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Οι ελεύθερε συναλλαγέ αποτελούν ακρηγονέο λίθο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται σαφήνεια βέβαια και το ξέρουμε αυτό και στην ε, Βρετανική και Ιρλανδική αγορά. Εμεί στην Ιρλανδία θέλουμε να έχουμε τέτοιε σχέσει. Η Αυστραλία με την Ιαπωνία και την Κίνα ήταν εμπορικό εταίρο μα το 2015 από του πιο μεγάλου με 2,5 δισεκατομμύρια. Υπάρχει μεγάλη παράδοση στις σχέσεις της Ιρλανδίας με την Αυστραλία και πολλοί Αυστραλοί προέρχονται από την Ιρλανδία ουσιαστικά. Οι σχέσει αυτές λοιπόν πρέπει να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο και αυτό προ το αμοιβαίο όφελο και των δύο πλευρών. Εκφράστηκαν διάφορε ανησυχίε για αρνητικέ συνέπειες μια τέτοια εμπορική συμφωνία στι δικέ μας ε, εξαγωγέ τροφίμων. Οι ανησυχίε αυτές είναι κάτι που παίρνω πάρα πολύ στα σοβαρά. Όντω ο αγροτροφικός τομέας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για μα. Και γι' αυτό και τις ανησυχίες αυτές πρέπει να τις λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Να υπάρξει μια ρήτρα αναθεώρησης ανάλογα με το πώς θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία. Ευχαριστούμε τελευταίως για αυτό την έκθεση ο κύριος Και Ένα λεπτό. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, εγώ στήριξα την έκθεση αυτή, η οποία έχει να κάνει με την διαπραγματευτική εντολή με την Αυστραλία. Πιστεύω ότι ακριβώ επειδή θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ελεύθερε συναλλαγές μα έχουν να χάσουν πολλά και ε, ξέρουμε ότι αυτό το θέμα αποτελεί ακρογωνία ολίθο για μα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσει πρέπει να αρχίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα και να εμείνουμε στι αρμοδιότητε μα και μόνο. Ευχαριστούμε. Περνάμε στην επόμενη έκθεση πάλι του κυρίου Κάσπαρη. Πρόκειται για διαπραγματευτική εντολή για εμπορικέ διαπραγματεύσει με τη Νέα Ζηλανδία. Ο κύριο Σελίμοβιτ έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν μετρήσουμε το μερίδιο της αγοράς για την Αυστραλία, για τις ειδικές επιχειρήσεις, αυτό το μερίδιο είναι τεράστιο και μπορεί να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Η εμπορική συμφωνία, λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει. Θα ήθελα, συνεπώς, να έχουμε μια σύγχρονη συμφωνία που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία και που να είναι και κατανοητή από όλους. Ευχαριστούμε. Σε ένα λεπτό καταφέρατε να μιλήσετε και για τις δύο τελικά συμφωνίες. Και εσείς για το ίδιο θέμα και και ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, στήριξα την έκθεση αυτή του κύριου Κασπάρη για τους ίδιους λόγους που τα έκανα και για την προηγούμενη έκθεση. Πρόκειται για μια έκθεση για διαπραγματευτική εντολή, εμπορικέ ε, διαπραγματεύσει με τη Νέα Ζηλανδία. Χρειάζεται νέε αγορέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται ελεύθερε συναλλογέ, γιατί αυτέ αποτελούν και το βάθρο ε, διαπραγματεύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να αρχίσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα, να τηρήσουμε και να σεβαστούμε τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στην περίπτωση της Αυστραλία όσο και στην περίπτωση τη Νέα Ζηλανδία που και οι δύο χώρε είναι σημαντικοί εμπορικοί εταίροι μα. Ευχαριστούμε και τελευταίος ο μιλητής τώρα, με τον οποίο έκλεισε η συζήτηση, ήταν ακριβώς αυτός. Α, κύριε και εσείς είσαστε... Α, τυχερός είσαστε, γιατί δεν τέλειωσατε η πρότασή μου με την οποία έκλεινα την ε, συνεδρίαση αυτή. Καλά. Τότε περνάμε στην τελευταία μας έκθεση για σήμερα που είναι ο έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο μόνος μας ο ομιλητής είναι ο κύριος Μάμικιντς. Ένα λεπτό. Λοιπόν, πάρτε βαθιά ανάσα και αρχίστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλές παραβάσεις γίνονται ακόμα και το τέλος του 2015 είχαμε 1.368 τέτοιες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου στον τομέα της απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων, περιβάλλον, δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα, εσωτερική αγορά, μεταφορές, υγεία, ε, πολιτισμός και εκπαίδευση. Κάθε καθυστέρηση είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και κάθε τέτοια παραβίαση γιατί πλήττει τις ζωές των ανθρώπων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει και ηλικέ επιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν στο μέλλον θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Κυβερνήσεις και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να κατανοήσουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, ποια είναι η πραγματική φύση των παραβιάσεων αυτών και μόνο τότε θα είμαστε σε θέση να τις αντιμετωπίσουμε και αποτελεσματικά. Υπερψήφισα. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε αγαπητοί συνάδελφοι. Ήταν τώρα πράγματι ο τελευταίος ο μιλητής. Έληξε η συνεδρίαση μέχρι τις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ.